το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στην πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Οκονή. Περατώθηκε η συζήτηση, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Τώρα, στην ημερήσια διάταξή μας, έχουμε την έκθεση Φλότ όσον αφορά την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων από την CIA σε ευρωπαϊκές χώρες. Δίνω το λόγο στην κυρία Φλότρα το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτούς τους εννέα μήνες που διήρκησε η εργασία μου, χάρη στη στήριξη και την εμπιστοσύνη, την ανεκτήμητη από όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία και κυρίως των Ευρωπαίων βουλευτών, οι οποίοι ποτέ δεν παρετήθηκαν από αυτή τη μάχη για τη δικαιοσύνη και για την αλήθεια, μετά από εννέα μήνες μπορέσαμε λοιπόν ε, να συγκεντρώσουμε επιβαρυντικά στοιχεία ε, για την Ευρώπη και τα κράτη της ως προς το μυστικό ε, πρόγραμμα της CIA. Οι έρευνε του Συμβουλίου τη Ευρώπη, η Ειδική Απεσταλμένη των Μένων Εθνών, ο Ερυθρό Σταυρό, οι ε, Εθνικέ Οργανώσει Υπεράσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουμε μαρτυρίες θυμάτων, των δικηγόρων του, αλλά και ε, πρακτόρων τη CIA. Ε, για όλα αυτά, σε όλους αυτούς πρέπει τα κράτη-μέλη να λογοδοτήσουν για ε, παθητική στάση ή για ε, πιο ενεργητική ε, κατάσταση σε, όλες αυτές τις, σε όλα αυτά τα βασανιστήρια που έχουν γίνει τα κράτη-μέλη έχουν επιδείξει αιμονή να καλύψουν την αλήθεια, έχουν επιδείξει πλήρη απουσία πολιτικής βούλησης, έχουν πρημοδοτήσει τα εθνικά συμφέροντα, έχουν προβεί ε, σε καταχρηστική ε, χρήση του δικαιώματος εθνικού απορρίτου και μυστικού έχουν ε, επιδείξει φοβερή φαντασία στους νομικούς τους συμβούλους και έχουν προβάλει με τελείως υπερβολικό τρόπο όλα αυτά τα εθνικά σύμβολα προκειμένου να μην χυθεί φως στην αλήθεια. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η έκθεση αυτή ώστε να ε, φανεί η στρατηγική των κρατών μελών η οποία είναι επίσημη τελικά τα τελευταία 11 χρόνια. Με τις συστάσεις στα κράτη-μέλη, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή η έκθεση εκφράζει τη σαφέστατη πολιτική βούληση να αξιοποιηθούν τα πάντα ώστε αυστηρές, ανεξάρτητες, διαφανείς έρευνες να γίνουν και να γίνονται ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη ε, στα θύματα και στις οικογένειές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη το χρωστούν αυτό στα θύματα αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι απαιτούν από όλα τα θεσμικά όργανα την τήρηση και τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών ε, που διέπουν το κράτος δικαίου που έχουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι ε, και έχουμε γίνει συγκεκριμένοι στην έκθεση. Μιλούμε για γεγονότα ώστε ε, τελικά να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα των μυστικών φυλακών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία από την Eurocontrol, την οποία ευχαριστώ. Είχαμε επισκέψεις από τους βουλευτές της Επιτροπής Πολιτικών Φιλελευθεριών και χάρη σε όλα αυτά ε, η έκθεση περιλαμβάνει πολύ ε, συγκεκριμένες συστάσεις ε, προς διάφορα κράτη-μέλη όπως η Πολωνία, η Λουθουανία και η Ρουμανία ε, τρεις χώρες που κατηγορούνται για βασανιστήρια και για μυστικά ε, κρατητήρια και φυλακές. Πρέπει να έχουμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση, ούτω ώστε να σπάσει πια αυτός ο νόμος της σιωπής. Το Συμβούλιο θα πρέπει επισήμω να επιληφθεί του θέματο, να το συμπεριλάβει στην ημερήσια του διάταξη, να αναγνωρίσει την ευθύνη που του αναλογεί και να απολογηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαπιστώσει τα γεγονότα. Αυτό όντω το έχει κάνει, αλλά δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει όλου του πόρου και όλα τα εργαλεία που έχει σε θέματα δικαιοσύνη και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να πιέσει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τι βασικέ υποχρεώσει του. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε πράγματι να εφαρμοστεί η αρχή αμοιβαία στήριξη και αλληλεγγύη. Κυρία Ρέντιν, η έκθοση μας κάνει να ε, σα δώσουμε ραντεβού, να σα καλέσουμε εσάς, να δώσουμε ραντεβού σε εσά, στο Συμβούλιο, στι οικογένειε των θυμάτων, ε, του χρόνου, σε ένα χρόνο. Την περασμένη εβδομάδα ένας Τούρκος ε, πολίτης, ο οποίος κρατεί το στη Γερμανία χωρίς δίκη και πριν πέντε χρόνια στο Γουαντάναμο χωρίς δίκη, ήρθε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας ε, διηγηθεί τον εφιάλτη του, τον Γολγοθά που έχει ε, περάσει. Ο κύριος Γκουρνάτς λοιπόν, εάν τον κρατήσουν οι δυνάμεις του και καταφέρει να έρθει πάλι του χρόνου να μας δει, τι θα πρέπει να του πούμε. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να να του απολογηθούμε εξ ονόμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του δείξουμε σε ένα χρόνο από τώρα αν καταφέρει να έρθει ότι πράγματι έχουν γίνει βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου προσωπικά να ευχαριστήσω την κυρία Φλότρο για τον τρόπο και το θάρρος με τον οποίο εργάστηκε και που ανέλαβε αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα άκρο ευαίσθητο. Είναι επίσης ένα θέμα που αφορά αξίες, τις αξίες μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα τόνισε ότι οι πρακτικές που αναφέρονται ως επιδόσεις, σε επιδόσεις, αποτελούν σοβαρή παραβίαση αρκετών θεμελιωδών δικαιωμάτων, παράνομη σύλληψη, αυθαίρετη κράτηση, βασανιστήρια, κακομεταχείριση. Και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές. Ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα τόνιζε ότι τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται όχι μόνο θα έπρεπε να σχολιάσουν, αλλά να διεξαγάγουν εις βάθος έρευνες για να λάμψει αλήθεια. Και αυτή είναι θετική υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ούτω ώστε να απαγγελθούν οι διάφορες ευθύνες και να μπορέσουν ε, να λάβουν αποζημιώσεις στα διάφορα θύματα για τις βλάβες και ζημίες. Και γι' αυτό αναφερθήκατε στο δικαστήριο, το οποίο ε, επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων. Από το 2005, όταν πρώτα ακούστηκαν αυτές οι εικασίες, η Κομισιόν είναι σε επαφή με εκείνα τα κράτη-μέλη ε, για τα οποία ακούστηκε πως είχαν μυστικά κέντρα κράτησης όσον αφορά την ε, πτυχή της αεροπορικής πολιτικής. Η Κομισιόν άντλησε τα διδαγματά της και υπήρξε σχετική ανακοίνωση για την πολιτική αεροπορία τον ε, Ιανουάριο του 2008 και βεβαίως υπάρχουν νέοι κανόνες για τα σχέδια πτήσης στον ενιαίο ουρανό οι οποίοι τέθησαν ενισχύ 1η 2009 και υπάρχουν νέα μέσα παρακολούθησης της πραγματικής κίνησης του αεροσκάφους και βεβαίως ε, Μπορώ να σα πω πω οι επαφέ με τα θεσμικά όργανα επί του θέματος είναι πάρα πολύ θετικέ. Επίσης η έκθεση αναφέρεται στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της ε, συμμόρφωσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία επί ποινικών ζητημάτων. Επ' αυτού η Κομισιόν είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει πω τα κράτη-μέλη θα ε, χρησιμοποιούν κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών μέσων και θα ε, συμμορφώνται με την χάρτα θεμελιωδών συγχωρείτε δικαιωμάτων. Γιατί, το έχω ήδη πει, ρητός ενώπιον του Κοινοβουλίου, πως ε, είναι ένα και το ευρωπαϊκό δίκαιο που ισχύει και στην περίπτωση αυτή είναι η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οπότε ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό αφορά όχι μόνο τις εσωτερικές στοιχές της δικαστικής συνεργασία, αλλά και τις εξωτερικές. Ως ε, προς αυτό η Κομισιόν τονίζει την σημασία ενισχύ ενισχύει από 1η Πρώτου 2010 των δύο συμφωνιών με τις ΗΠΑ για την έκδοση και την αμοιβαία νομική αρρωγή. Και οι δύο ξεκαθαρίζουν και ενοποιούν το νομικό πλαίσιο δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά ζητήματα με τις ΗΠΑ και αναφέρονται ρητός στην ανάγκη ε, πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τις εθνικές και θεσμικές ελλείψεις που τόνισε η έκθεση. Να υπενθυμίσω πως οι υφιστάμενες συνθήκες δεν δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συστήσει ένα γενικό μηχανισμό για τις παραβιάσεις των θεμελιών δικαιωμάτων. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η Κομισιόν επαγρυπνεί για να διασφαλίσει πως ο χάρτης ισχύει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου όπως εξήγησα για την συνεργασία σε ποινικά ζητήματα. Όσον αφορά τώρα την υποπτία των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών. Ξέρετε πως είναι μια, ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Κομισιόν έχει επαναλάβει πως η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να καταστρατηγεί τα σχετικά ευρωπαϊκά μέσα στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικά δήματα. Καμία συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών δεν μπορεί να υπονομεύσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου. Και νομίζω πως το Κοινοβούλιο συμφωνεί μαζί μου και αυτό είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την τρομοκρατία. Όταν εφαρμόζουμε δηλαδή τους βασικούς κανόνες επί των οποίων οικονομήθηκε η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεργαστεί ενεργά με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε αυτό το οποίο συνέβη στο πλαίσιο των λεγόμενων παραδόσεων ανθρώπων στη CIA να μην ξανασυμβεί ποτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Το λόγο έχει τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων η συνάδελφος κυρία Λάτφορτ Σάρα. Για δύο λεπτά. E Πρόεδρε, έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει δημοκρατία και κάτω δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αξιόπιστες εικασίες για τη συνεργασία με τη ΑΕΕ για παράνομες παραδόσεις και κρατήσεις και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Ε, κάτι πολύ κακό. Αλλά αυξάνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει συνεργασία στη διερεύνηση των γεγονότων. Κολυσιεργία όσον αφορά τι έρευνε, τι εθνικέ και τι διεθνεί, είναι κάτι που ντροπιάζουν την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Ε, να θεωρείται κρατικό μυστικό και να διονύζεται τιμωρησία είναι κάτι απαράδεκτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει το κουράγιο και να μπορέσει να ελέγξει το κατά πόσο τα κράτη-μέλη έχουν συμμετάσχει τις πράξεις. Διορίσαμε τον Σταύρο Λεμνινίδη, ο οποίος είναι ο πρώτος υπεύθυνός μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει σε όλο τον κόσμο ε, να γίνονται σεβαστά ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά υπονομεύεται αυτό από το γεγονός ότι υπάρχουν υπόνοιες ότι κάποια κράτη-μέλη μπορεί να συνεργάστηκαν με τη CIA για αυτές τις πράξεις. Θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις αξίες μας, τις εξωτερικές μας σχέσεις. Δεν είναι μόνο μια αρχή, είναι αναγκαίο. Κοιτάξτε γιατί στη Λιβύη. Υποτίθεται ότι βασανίστηκαν με τη συνεργασία δυτικών κυβερνήσεων άνθρωποι και των μυστικών υπηρεσιών και αυτοί που είχαν συνεργαστεί είναι τώρα στην κυβέρνηση που ακολούθησε τον Καντάφη και ο Τόνι Μπλερ θα πρέπει να δικαιολογηθεί και αυτό και ο Τζορτζ Μπούς ο οποίος δημιούργησε ε, ουσιαστικά το χώρο του κατάναμου και δεν σεβάστηκαν ούτε οι δημοκράτες πρόεδροι το δίκαιο μας απογοήτευσε και ο πρόεδρος ε, Ομπάμα δεν έκλεισε τον Κατάναμο ούτε ρίξε φως στο παρελθόν και επιμένει να υπάρχουν στρατιωτικές επιτροπές που επιβάλλουν θανατική ποινή, τα στατοδικεία. Και επίσης και γίνονται δολοφονίες με μη επανδρομένα επτάμενα οχήματα. Θα πρέπει να α, θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη ακόμα μετά από δεκαετίες. Θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να ρίξουν φως στην φρικτή αυτή περίοδο υποστηρίζοντας τους ειδικούς ε, εισηγητές και ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών στο έργο αυτό. Ευχαριστώ. Ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η, κυρία, η συνάδελφος κυρία Μισελ Στρίφλερ για δύο λεπτά. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επιτρόπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάθε μέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να κάνουμε το πάνω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι να είναι ένας χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, να είμαστε όσο δυνατόν πιο κοντά στο πολίτη ε, και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος όπου θα πρέπει να επικρατεί και να υπερισχύει, υπερισχύει το κράτος δικαίου και όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να χαίρουν προστασίας. Αυτές είναι οι αρχές που μας διέπουν, εμένα προσωπικά αλλά και την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκω. Ε, κύριε Πρόεδρε, αύριο είναι η δέκατη η επέτειος από την επίθεση στο World Trade Center στη Νέα Υόρκη η Ευρώπη πάντοτε ε, συνεχίζει να διαβεί υπό την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων. Ισχύουν και επιμένουν οι τρομοκρατικές ε, επιθέσεις, υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ο οποίος επιμένει και δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Επομένως, θα πρέπει ε, να έχουμε αντιτρομοκρατική πολιτική που να βασίζεται στους σωστούς πυλώνες, δηλαδή ε, στο κράτος δικαίου και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα δύο αυτά δεν είναι αντιφατικά μεταξύ τους, είναι άλληλο συμπληρωματικά. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, μυστικές κρατήσεις χωρίς απαγγελία κατηγοριών, χωρίς διεξαγωγή δίκης είναι πράγματα που αντίκειται, ε, αντίκειται στις δικές μας αξίες και δεν πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό χώρο. Κανείς δεν μπορεί να μην έχει, να του αρνηθούμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και πρέπει να εγγυόμαστε την δίκαιη δίκη σε όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια εξ ονόματος της ομάδος είναι η συνάδελφος κυρία Τάνια Φαγιόν για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν κάποιοι ακόμα αναρωτιούνται γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από όλα αυτά τα χρόνια ακόμα ασχολείται με το ζήτημα των παράνομων απαγωγών κρατήσεων και βασανισμών των ανθρώπων αυτών σε ευρωπαϊκό εφόσον Να σας υπενθυμίσω πως η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βεβαίως δεν παραγράφεται. Η ε, δουλειά αυτή δεν ήταν εύκολη, δεν ήθελαν τα κράτη-μέλη να μας δώσουν δεδομένα, μιλούσαν για κρατικά μυστικά. Αύριο λοιπόν θα δώσουμε την ικανοποίηση στους ανθρώπους αυτούς της προειδοποίησης των οποίων αγνοήσαμε για χρόνια και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε όλους αυτούς οι οποίοι υπέφεραν λόγω της πολιτικής που προέκυψε από τα γεγονότα αυτά που έγιναν πριν από μία δεκαετία. Και μην ξεχνάμε πως κανένα κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί ακόμα πλήρως με τις υποχρεώσεις του για την ε, πρόστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις διεθνείς διαδικασίες ε, για την αποδόση ευθυνών στα κράτη-μέλη μόνο. Έτσι θα μπορέσουμε να εκτίσουμε την φήμη μας για ε, την διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μόνο έτσι θα μπορούμε σοβαρά να απαιτούμε από υποψηφίες χώρες και χώρες στη γειτονιά μας να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική νομιτάξη. Ευχαριστώ. Στο βήμα εξ της των η συνάδελφος κυρία Σοφία Ινετβέλτ για δύο λεπτά. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω λέγοντας πως ε, όπως ε, τόσο συχνά στις ε, συζητήσεις αυτές αποσιάζει το Συμβουλίο. Από ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα και εξ ονοματός τους. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την εισηγήτρια η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε άρνηση και ε, όταν ακούω τους συναδέλφους του ΕΛΚ φαίνεται πως και το ΕΛΚ βρίσκεται σε άρνηση. Αυτό το οποίο είναι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εάν τα ίδια πράγματα τα είχαν κάνει άλλες χώρες, π.χ. αραβικές, ε, θα ήταν γεμάτη αίθουσα. Θα ήταν εδώ το Συμβούλιο. Και πάρα πολύ γρήγορα θα καταδικάζαμε αυτές τις πράξεις. Αλλά επειδή έγιναν με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, δεν θεωρούμε πως πρέπει να δώσουμε λόγο σε κανέναν. Έχουμε χάσει εδώ πέρα το ηθικό μας έρισμα και την αξιοπιστία μας και είναι τραγική η ηρωνία στο ότι βοηθούμε εμείς να εκτοπίσουμε δικτάτορες όπως ο Καντάφη, ο Μουμπάρακ, ο κύριος Ασάντ που ακόμα κυβερνάει που ήταν σύμμαχοί μας μέχρι πρότινος και λέμε σε αυτές τις χώρες, ε, στη χώρα του κυρίου Ασάντ, ε, τους στέλνουμε ανθρώπους γιατί είναι τόσο καλή στα βασανιστήρια. Ε, είναι έσχος την σήμερα ημέρα ακόμα να μην απαντούν οι κυβερνήσεις της Ευρώπης να παραδεχτούν τις ευθύνες τους και να ζητήσουν συγγνώμη. Συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι η μία ή η άλλη χώρα. Είναι συλλογική η ευθύνη. Το θέμα δεν αφορά τη Ρουμανία, τη Λιθουανία ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε μία κοινότητα αξιών και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε καθήκον. Δεν θα ξεχάσουμε, θα συνεχίσουμε να φύγουμε αυτό το θέμα μέχρι κάποιοι να λογοδοτήσουν για ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγιναν εξ ονόματός μας. όνομα της ομάδας των Πρασίνων, ε, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Φρίντα Μπρέπελς για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ήμουν ε, τότε μέλος της Προσωρινής Επιτροπής για τη CIA στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως θα ήθελα να συγχαρώ εξ ονόματος ομάδας μας ε, και την ε, εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Γιατί στον καιρό της έκθεσης ε, Φάβα ήταν πάρα πολύ συνάδελφο να... ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε το τι γίνεται. Δεν υπήρχαν πληροφορίες για το πρόγραμμα απαγωγών και κρατήσεων της CIA. Και ακριβώς εδώ πέρα βρίσκεται η δύναμη αυτής της έκθεσης, συγκεκριμένες πληροφορίες και στις συστάσεις δηλαδή. Καθώς ε, επίσης ε, και στο ότι το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει επαρκής ορισμός της ε, τρομοκρατίας, καθώς και δημοκρατικός έλεγχος των υπηρεσιών πληροφοριών. Οπότε μιλάμε για απαγωγές και αυθαίρετες κρατήσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον. Αυτά λέγαμε τότε, πριν από πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια μετά βλέπουμε πως όλα αυτά έμειναν κενό γράμμα και δεν έχει υπάρξει απολογισμό σε διάφορα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατόν να παραμένει κουφή σε αυτά τα οποία ακούγονται για τη δική της εμπλοκή στο πρόγραμμα της CIA και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΗΕ, τα ΜΜΕ και οργανώσεις όπως η Εθνική Αμνηστία ασχολούνται με το θέμα. Ελπίζω πως το Κοινοβούλιο μετά από αυτήν την έκθεση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση μέχρι να καταλήξουμε στο να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις συστάσεις. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο γιατί οι αυθαίρετες κρατήσεις δεν έχουν ακόμα τελειώσει, ειδικά στις ΗΠΑ και παρόλες υποσχέσεις δεν έχει κλείσει το Γουανταναμό. Βεβαίω είναι αναγκαία η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει παραβίαση των προσωπικών ελευθεριών. Αυτό είναι απολύτως σημαντικό για όλους και θα πρέπει η ευρωπαϊκή αντιδρομοκρατική πολιτική να μπορεί να ε, διασφαλίσει και να διαβεβαιώσει πως υπάρχει ένα δημοκρατικό πλαίσιο, πλαίσιο λειτουργίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως με το να συνεργάζεται χωρίς καμία κριτική η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα της CIA, με το να δίνονται διπλωματικές διαβεβαιώσεις και ο τρόπος με τον οποίο οι υπηρεσίες ε, πληροφοριών έπαιξαν αυτό το παιχνίδι, έπληξαν τα θεμέλια της Ευρώπης, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ομάδα μου είναι υπέρ και ενός πιο έντονου κειμένου που θα καταδικάζει αυτές τις πρακτικές για να διατηρήσει το ηθικό της αίρισμα η Ευρώπη στον κόσμο. Ευχαριστώ. συνάδελφε, on behalf of the ECR, ε, I will now give the floor του... Τώρα δίνουμε το λόγο στον συνάδελφο Τίμωθη Κέρκοπ για το ECR για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, και εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Οι ισχυρισμοί για την εμπλοκή ορισμένων κρατών μελών πρέπει να εξεταστούν με απόλυτη σοβαρότητα και να γίνει έρευνα σε βάθος. Ως νομικός, ως δημοκράτης και ως πρώην Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων πιστεύω ότι ε, τέτοια έρευνα πρέπει να γίνει μέσω μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας, ε, μέσω ανεξάρτητης ε, ανακριτικής διαδικασίας η οποία ενδεχομένω έχει ήδη και ξεκινήσει ε, στις ενδιαφερόμενες χώρες. Ε, θα πρέπει να κάνουμε το πάνε για να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ε, πραγματικές αποδείξεις, είτε αθωωτικές είτε καταδικαστικές. Εάν δεν τα καταφέρνουμε αυτά, με τέτοιου είδους εκθέσεις ουσιαστικά προσφέρουμε βοήθεια σε όσους θέλουν να προπαγανδίσουν και ε, σε διάφορες ομάδες. Εγώ ε, θέλω να υπάρχει έρευνα ούτως ώστε να αποκατασταθεί η φήμη των υπηρεσιών ε, που έχουμε για την ασφάλεια, των υπηρεσιών πληροφόρησης, διότι πιστεύω ότι έχει λερωθεί το όνομά τους αυτή τη στιγμή. δακτυλοδείχνονται και άλλα κράτη-μέλη. Κατηγορούνται αλλά δεν καταδικάζονται. Είναι δίκαιο αυτό. Βεβαίω και είναι σημαντικό να συνεργαστούμε περισσότερο, να διασφαλίσουμε μια καλή μεθοδό εργασία ε, για την ε, ε, συμφωνία για αυτό το ψήφισμα. Ωστόσο, το περιεχόμενο, η γλώσσα, η διατύπωση αυτή τη έκθεση, αλλά και η προσέγγιση που υιοθετεί το πνεύμα τη δεν μας βοηθά να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Εγώ έρχομαι από μια χώρα, κύριε Πρόεδρε, όπου πράγματι κανείς είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν αρκεί σε κάποιους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, Γκουε, το λόγο έχει κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι προς τιμήν μας. Ε, και ο τύπος και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις το έχουν επισημαίνει επανειλημμένος. Μυστικές επιχειρήσεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου έγιναν από τη CIA με την εμπλοκή και συμμετοχή πολλών κρατών σε όλο τον κόσμο και τελικά είχαμε απαγωγές, εξαφανίσεις, βασανιστήρια ε, διαφόρων ενδυνάμει υπόπτων και διοχέτευσή τους προς το Γουαντάναμο το οποίο δυστυχώς δεν έχει κλείσει ακόμα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη έκαναν τα πάντα και συνεχίζουν να το κάνουν ορισμένα από αυτά προκειμένου να αποκρύψουν ε, την αλήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου την εισηγήτρια, την κυρία ε, ε, Φλότχο διότι έκανε αυτό το αυτή τη πάρα πολύ δύσκολη δουλειά παρά τα εμπόδια στα οποία προσέκρουε συνεχώς. Θέλω να πω ότι Κανείς δεν παραδέχεται ότι αλλάζει την οπτική του γωνία και την ανάλυση που κάνει αναλόγως ε, με το αν είναι συμπολίτευση ή αντιπολίτευση στη χώρα του. Αυτό πρέπει όμως να το ομολογούμε. Και ε, καλό θα είναι να διδαχθούμε από κράτη που πραγματικά έχουν ε, διδάξει τα υπόλοιπα. Κανένα κράτος, είτε είναι η ΕΠΑ, είτε είναι κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να απεκδηθεί των ευθυνών του, ειδικότερα όσον αφορά ε, την καταπολέμηση της, αξιο... της τρομοκρατίας. Ναι, είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι ενώπιον των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε. Και θα πρέπει πρώτα η Ευρώπη να καθαρίσει τα του οίκο τη και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Ε, Δίνω τον λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Ανδρέα Μέλτσερ για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο διδάσκει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μακρινές χώρες και απειλεί με κυρώσεις. Και βεβαίω αυτό είναι κάτι στο οποίο δεσμεύονται όλες οι υποψήφιες χώρες μέσω της ΕΣΔΑ όπω ξέρουμε και είναι σκάνδαλο με δεδομένα αυτά πως ε, συμμετείχαν ε, κάποιες ε, χώρες σε παράνομες μεταφορές κρατωμένων και συζητήσεις της CIA και από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε μόνο γνώση αλλά και συνέργεια εθνικών κυβερνήσεων και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Σαν να μην έφτανε δε αυτή η παραβίαση της ΕΣΔΑ έχουμε και τις ατελείωτες καθυστερήσεις. Έχει φτάσει η ώρα επιτέλους να κάνουμε κάτι και να κλείσει αυτή η υπόθεση. Όταν όμως μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως ειδικά α, καθώς έχουμε τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο τι συμβαίνει εκεί πέρα. Μόνο και αυτή η συμφωνία με τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης κατά την άποψή μου αρκεί για να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να μιλήσουμε για μια προνομιακή σχέση. Και αν μιλάμε σοβαρά για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να δούμε και ιστορικούς ε, νόμους ε, που ήταν άδικοι όπως παραδείγματο χάρη η Σλοβενική ή τα διατάγματα Μπένες στην Τσεχοσλοβακία τότε. Ευχαριστώ. Το λόγο στον συνάδελφο κύριο Κάρλος Κοέλιο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αγαπητή κυρία Επίτροπε, ο κύριος Φρατίνη είπε ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να επιτυγχάνεται με κάθε τίμημα. Το έχει δηλώσει αυτό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης έχει γίνει αναφορά ε, στο τεκμήριο της αθωότητας ενώπιον ανεξάρτητου ε, δικαστηρίου ε, και έχει γίνει αναφορά και στο δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Τα λέμε όλα αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει για τους ανθρώπους που διαβιούν στο Γουαντάναμο. Στην έκθεση που έχω μειοθετήσει στις 14 Φεβρουαρίου του 2007, εξετάσαμε όλα αυτά τα γεγονότα και βρήκαμε στοιχεία πολύ επιβαρυντικά, παραλήψεις, ε, κάναμε συστάσεις και θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί αυτές οι συστάσεις για να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα. Τι θα γινόταν αν τέτοιου είδου πράγματα συνέβαιναν σήμερα. Θα ήταν η ιστορία διαφορετική, ο κόσμος θα αντιδρούσε διαφορετικά. Εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν θα γινόταν. Μια από τα ίδια θα είχαμε. Ενδεχομένω ο κόσμο γνωρίζει περισσότερα, τα μέλη του Κοινοβουλίου ε, είναι σε ένα στάδιο έτσι περισσότερη εγρήγορση και ορισμένοι ενδεχομένω θα αντιδρούσαν πιο γρήγορα. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, και οι κυβερνήσει των κρατών μελών δεν κοίταξαν τι 40 συστάσει που είχαμε κάνει στην έκθεση τότε πριν από αρκετά χρόνια. Εγώ στηρίζω τι συστάσει σα. Οφείλω όμω να πω ότι αυτό που αναφέρεται για λόγους έκτακτης ανάγκης του κράτους ε, θα πρέπει να γίνεται πάρα πολύ καταξαίρεση και να μην χρησιμεύει ως χιτώνας κάλυψης πραγμάτων που δεν θα όφυλαν και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδου ασυλία. Οφείλουμε να συνεργαστούμε στενά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών, ώστε οι 40 συστάσεις που έχουμε εμείς εγκρίνει στο παρελθόν να εξεταστούν μία προς μία και να εφαρμοστούν κιόλα. Η... Ενδεχομένως είναι δύσκολο αυτό, ωστόσο ε, πολύ λίγα έχουν εφαρμοστεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Έχει τώρα η συνάδελφος κυρία Σιλβή Γκυγιόμ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, όπως και οι συνάδελφοί μου, συγχαίρω και εγώ τη συνάδελφο και η κυρία Φλότχο για τη δουλειά που έκανε και τι προσπάθειε που κατέβαλε, ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν τους όλες οι αρχές ε, σε αυτό το πολύ τοπίο αυτής τη υποθέσεως έχουν παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλέ χώρε επί ευρωπαϊκού εδάφου και έχουν περισσότερε ερωτήσει από απαντήσει. Η καταπολέμηση τη τρομοκρατία δεν μπορεί να δικαιολογεί τα πάντα, διότι έτσι χάνει κάθε νομιμότητα. Θα ήθελα να επιμείνω ε, τι τάσει επί τη κατάχρηση τη αρχή του κρατικού μυστικού ή του εθνικού μυστικού. Είναι ένα εμπόδιο στον αφορά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα πρέπει και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα ευρωπαικα κράτη-μέλη να επιβάλλουν τη διαφάνεια έτσι να αποκασταθεί η αξιοπιστία όσον αφορά το δημόσιο τομέα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σεβόμενοι όλοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα κάποιε χώρε, αλλά υπάρχει συλλογική ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα πρέπει να τοποθετήσει σαφώ το Συμβούλιο επί των οικασιών και των συγκεκριμένων γεγονότων όσον αφορά τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να αποσιοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άλλη θα πρέπει να αξιολογήσει ε, σύμφωνα με τις συνθήκες αυτά που έγιναν και να ρηχθεί άπλο το φως στην υπόθεση. Δράτω με τις ευκαιρίες για να συγχαρώ τους πολίτες που κινητοποιήθηκαν και είναι πολύ άριθμοι όσον αφορά αυτή την έκθεση και περιμένω υπόμονα την ψηφοφορία ούτω ώστε κάτι να κινηθεί επιτέλους και ελπίζω ότι αύριο θα υπάρξει μεγάλη υποστήριξη από πλευρά Κοινοβουλίου στον αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε το λόγο έχει τώρα κύριος Κόνραντ Σιμάνσκι για ένα λεπτό. Dziękuję Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα μισά κράτη-μέλη διέθεσαν τον ενέργειο χώρο τους για τις πτήσεις της CIA. Σημαίνει αυτό πως τα μισά κράτη-μέλη αμέλησαν ε, ε, να προστατεύσουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική παράδοση του διεθνούς δικαίου δεν νομίζω πως ε, είναι αυτό το σωστό συμπέρασμα. Νομίζω πως ε, τα κρατη αυτά έλαβαν δύσκολες αποφάσεις και δεν υπάρχει εμφιβολία πως έγιναν λάθη. Αλλά θα ήταν υποκριτικό να κατηγορήσουμε τα μισά κράτη-μέλη χωρίς μια εναλλακτική για το τι πρέπει να γίνει με ε, το στελέχη της Διεθνούς Τρομοκρατίας. Και η πρόταση να δοθούν στους τρομοκράτες τα ίδια δικαιώματα με οποιονδήποτε άλλον πολίτη δεν είναι σωστή. Και ο πρόεδρος Ομπάμα επίσης το αντιλήφθηκε αυτό. Και σήμερα η φυλακή του Γκουαντανάμου εξακολουθεί να λειτουργεί και ο πρόεδρος των ΙΠΑ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ε, στρατοδικία για να δικάσει ε, αυτούς τους τρομοκράτες. Αλλά δεν το αντιλαμβάνεται αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Κύριε Σιμάνσκι, η συνάδελφος κυρία Ινετβέλτ και ακολούθως η, κυρία, η συνάδελφος κυρία Λάτφορτ θέλω να κάνω χρήση της μπλε κάρτας. Κυρία Ινετβέλτ. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει η διερμηνία, αλλά μας είπε πράγματι ο κύριος Σιμάνσκι πως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ύποπτοι τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες. Απορρίπτεται δηλαδή την αρχή πως τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους και τι σημαίνει αυτό. Δεν ε, υποστηρίζετε και όλες τις αξίες που υπάρχουν στις ε, συνθήκες μας. Ευχαριστώ. E, Λέει λοιπόν ο Σιμάνσκι, ε, συμφωνώ με την αρχή των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά ο καθορισμό του εγκληματία, η κατάσταση για έναν εγκληματία είναι διαφορετική από κάποιον που ε, που, κάνει να εκραγεί μια βόμβα και είναι ένας τρομοκράτης. Και χρησιμοποιούνται διαφορετικές διαδικασίες για δύο διαφορετικές υποθέσεις. Έχουμε τα πολιτικά δικαστήρια και τα στατοδικεία. Οι τρομοκράτες δεν διαπράττουν απλά δικήματα, απλά εγκλήματα, αλλά διαπράττουν κάτι που μοιάζει με στατιωτικά εγκλήματα. Οπότε δεν μπορεί η πολιτική δικαιοσύνη να αντιταχθεί στα προβλήματα της τρομοκρατίας. Οπότε υπάρχει ένα νομικό κενό. Κύριε Σιμάνσκι, ενισχύεται την ανησυχία μου για το αρχικό σας σχόλιο. Επιμένω λέγοντας ότι τρομοκρατικές πράξεις είναι εγκλήματα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όπως τα άλλα εγκλήματα. Να δικάζονται, να υπάρχει δίκαιη δίκη το κάναμε με άλλα διεθνή εγκλήματα μέσα του Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου και το, ε, του, δικαστηρίου, του Ποινικού Δικαστηρίου. Αλλά μετά την 11η Σεπτεμβρίου ε, όλα υπονομεύθηκαν. Θα έπρεπε να συνεργαστούμε για να εφαρμόζεται το διεθνέ δίκαιο παντού και οι τρομοκράτε να δικάζονται. Κάτι που δεν έγινε σαν αντίδραση άμεση μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Σιμάνσκι, συμφωνώ ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφαίνεται σχετικά με τις ποινές που θα επιβάλλονται και στους απλούς εγκληματίες και στους εγκληματίες πολέμου και στους τρομοκράτες. Αλλά απλή νομική διαδικασία δεν αρκεί όταν θέλει να αντιμετωπίσει κανείς ένα τρομοκρατικό δίκτυο. Και η συνθήκη της Γενέβης, οι συμβάσεις της Γενέβης έχουν συνταχθεί εδώ και 60 χρόνια και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση. Και κυρίως, και κυρίως οι διάφορες ποινικέ διαδικασίες δεν μπορούν να το καλύψουν αυτό. για Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για παράνομη μεταφορά και κράτηση ανθρώπων και όλο αυτό δείχνει ε, ότι έχουμε ε, προληπτική αντίληψη για την πάταξη της τρομοκρατίας και όλα αυτά ε, υπάρχουν στο γλωσσάριο εντό εισαγωγικών που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ. Αυτό φαίνεται και έχει τύχει στήριξη από τα κράτη που έχουν αντιμετωπίσει τρομοκρατικές απειλές. Είναι μια έννοια ε, που επικαλέστηκε τον ΝΑΤΟ για να καταστρατηγήσει ανθρώπινα δικαιώματα ε, και να επιβάλλει τη βούλησή του. Όλα αυτά αναγνωρίζονται στην έκθεση Φλότχ και τελικά καταστρέφεται ένα πλαίσιο ειρηνικού διαλόγου και συμβίωσης το οποίο είχαμε καταφέρει να εδραιώσουμε και να θεσμοθετήσουμε στον ΟΗΕ από το 1945 μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά όλα αυτά ε, το μόνο που κάνουν είναι να πρημοδοτούν τις υπεριαλιστικές πολιτικές των ΙΠΑ και των ε, συμμάχων τους. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ερευνήσουν σημαντικά τα στοιχεία που υπάρχουν για την εμπλοκή τους ε, σε τέτοιου είδους πράξη. Στην Πορτογαλία κάναμε το παν για να υπάρξει τέτοιου είδους έρευνα η οποία θα επιρρύψει τις ευθύνες που τις αναλογούν στην κυβέρνηση ε, της εποχής. Δυστυχώς αυτή η διαδικασία ε, μπλοκαρίστηκε από τα ε, ε, εθνικιστικού χαρακτήρα κόμματα που έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο όμως. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σεβόμεν την ένωμη τάξη. Κυρία Έλενα Μπασέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε ε, όλο αυτό τον καιρό. Ως κοιόδη εισηγήτρια από πλευράς ΕΛΚ έχω συμβάλει στην ε, κατάρτιση της έκθεσης αυτής. Ανέκαθεν θέλησα το τελικό κείμενο να είναι αντικειμενικό, να είναι ισορροπημένο και να υπογραμμίζει τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει τα πέντε τελευταία χρόνια, εάν αυτά έχουν υπάρξει και όπου έχουν υπάρξει ταυτοχρόνως καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Ζήτησα και ζητούσα η έκθεση να μην αποτελεί καταγγελτήριο λόγο εναντίον των κρατών μελών μόνο, διότι δεν μπορεί ένα κοινοβούλιο να ε, καθιστά ε, τους μηχανισμούς σωστής διεξαγωγής, ανάκρισης και έρευνας σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο. Ένα κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι ε, δικαστήριο και να αποδώσει ευθύνε χωρίς να έχει υπάρξει πραγματική εξέταση και διερεύνηση της υπόθεσης. Θέλησα η έκθεση αυτή να εξηγεί με πιο ισορροπημένο τρόπο την κατάσταση στα διάφορα κρατημέλη συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας. Και χαίρομαι διότι η έκθεση παραπέμπει τελικά στην κοινοβουλευτική έρευνα του 2000 τόσο εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα μου την Ρουμανία. Είχαμε ίδια πρωτοβουλία για την έκθεση αυτή και είχε φανεί ότι είχε, ε, ε, έχει υπάρξει παραποιημένη εικόνα της πραγματικότητας και εν μεταξύ έχουν προκύψει και νέα στοιχεία. Ε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε, έχει σημασία αυτό, ότι ορισμένα στοιχεία που είχε παρουσιάσει ο τύπος τότε κατά κόρον τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Επομένως, κάθε αίτημα επιπρόσθετης έρευνας, για να γίνει επιπρόσθετη έρευνα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη νέων και αδιάσυστων στοιχείων. Το τεκμήριο της αθωότητας θα πρέπει πάντοτε να προστατεύεται. Άλλωστε τελικά ο σκοπός μας είναι να ε, βρούμε ποια είναι η αλήθεια και όχι να βρούμε ενόχους με κάθε τίμημα. Είναι ο συνάδελφος κύριος Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η έκθεση είναι κάτι απαραίτητο. Θέλουμε να διευκρινιστεί η κατάσταση όσον αφορά των εικαζόμενων κέντρων κράτησης της CIA στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το έγγραφο όμως γίνονται αναφορές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση. Η τελική έκθεση πρέπει να είναι αντικειμενική και να δείξει ποιες είναι δεχόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς, εδώ υπάρχουν κατηγορίες άμεσες που απευθύνονται κατά κάποιων κρατών μελών χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις. Άρα δεν θα μπορέσω να υποστηρίξω απόλυτα αυτή την έκθεση. Η έκθεση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι ήδη, να θεωρηθεί ότι ήδη γνώριζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχε αποδείξει και ήξερε ότι υπάρχουν αυτά τα κέντρα κρατήσεων τη CIA. Εμεί έχουμε σαν ρόλο να εκπροσωπούμε του Ευρωπαίου πολίτε. και όχι να αντικαταστήσουμε τι ειδικευμένε δικαστικέ αρχέ. Αυτέ οι αρχέ θα πρέπει να παίξουν τον ρόλο του, οι ένοχοι θα πρέπει να πληρώσουν και δεν θα πρέπει να επαναληφθούν ποτέ αυτά. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Σαγιάτ Καρίμ. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι πριν από 7, θυμάμαι ότι πριν 7 χρόνια στεχόμουν εδώ και η χώρα μου είχε την Προεδρία ε, και είχαμε θέσει τον κύριο Αλεξάνδρ ε, τότε για τις εικασίες που είχαν ε, εκφραστεί και άκουσα την ε, οργή του και την οργή του Υπουργού Εσωτερικών και έφυγα υπό με... γέλια από αυτήν την αίθουσα, με κορόιδευαν. Και σήμερα κύριε Πρόεδρε πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη σημαία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Μόνο δύο θεσμικά όργανα είναι εδώ και οι θέσει του Συμβουλίου είναι κενές, άρα υπάρχει έλλειψη αφοσίωση ή αναγνώριση από πλευρά των εθνικών μας κυβερνήσεων. Αν ήταν τρίτες χώρε οι που, τις οποίες αφορούσε αυτές οι εικασίες, αναρωτιέμαι τι αντίδραση είχαμε τότε. Στο Ενωμένο Βασίλειο βεβαίως τώρα έχουμε κάνει διαφορετικά βήματα. Έχουμε δική μας εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται απορρίπτοντας αυτά που θα είχαν γίνει πριν. Δεν αρκεί αυτό όμως. Όταν οι τρομοκράτες ε, κάνουν κάτι, δεν είμαστε αδύναμοι όταν διατηρούμε τις αρχές. Δεν μπορούν να μας καταστρέψουν μέσω των δράσεών, σας, τους, αλλά μπορούν να πάρουν πολλά μέσω των αντιδράσεών μας. Και τι λέω στον κύριο Σιμάνσκι όταν κάνει διάφορα εθνικιστικού τύπου σχόλια και φεύγει την αίθουσα. Να του πω ότι υπάρχει μια χώρα που δεν ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι και να μάθουμε πολλά. Και είναι η Νορβηγία. Όταν αντιμετώπισε την, τα πιο φρικτά εγκλήματα, βομβαρδισμούς και θανάτους δεν αντέδρασε αφαιρώντας τα δικαιώματα των πολιτών, έδωσε κάθε δικαίωμα και απέδωσε δικαιοσύνη. Και σήμερα θα πρέπει να χαιρετήσουμε την Ορβηγία για αυτό που έκανε. Ευχαριστώ πολύ, ε, συνάδελφε κύριε Καρύμ. Ανοίγει η διαδικασία Catch the και δίνω το λόγο ευθύ αμέσω στη συνάδελφο κυρία Φλάσκοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόγραμμα της ε, CIA είχε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφορούσε τις παραδόσεις CIA, εξαφανίσεις, βασανιστήρια. Υπάρχει μια ειδική επιτροπή που έρευνα ε, αυτά τα γεγονότα το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει συνεργασία των εθνικών κυβερνήσεων για το ζήτημα αυτό. Η Ένωσή μας βασίζεται στο σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιώδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις και τα λοιπά. Για να διατηρηθεί λοιπόν η πίστη των πολιτών μας και η εμπιστοσύνη του στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να ε, είμαστε υπεύθυνοι και στον τομέα της ασφάλειας. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να ερευνούν τις κατηγορίες αυτές, ακόμα δεν έχουν συμμορφωθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη ε, συχνά μιλάνε για δημοκρατικέ αξίε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμω η εμπλοκή πολλών ευρωπαϊκών κρατών σε κατάφορε παραβιάσει των βασικότερων δικαιωμάτων αποδεικνύει πω όλα αυτά τα λόγια είναι μόνο ρητορίε. Μιλάμε για συνέργεια σε κρατικέ απαγωγέ, εξοδικαστικέ φυλακίσει και βασανιστήρια. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και γνωστά στι εμπλεκόμενε κυβερνήσει στον Κουαντανάμο και όλα τα μυστικά κέντρα στην Ευρώπη πρέπει να κλείσουν αμέσω Όλοι οι κατηγορούμενοι πρέπει να πάνε σε δίκη ή να απελευθερωθούν. Πέρσι 20.000 ε, Αμερικανοί στρατιώτε πέρασαν από το αεροδρόμιο Σάνων στην Ιρλανδία και τουλάχιστον διευκόλυνε επίση το ίδιο αυτό αεροδρόμιο την ε, παράδοση αυτών των ανθρώπων. Ζητάω να ε, επιθεωρούνται όλα τα στρατιωτικά αεροσκάφη που περνάνε από το αεροδρόμιο Σαν και υπενθυμίζω στον κύριο Γκίλμορ και το εργατικό κόμμα τη θέση που είχαν στην αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η παράνομη κράτηση και ανάκριση που πραγματοποιεί η CIA είναι κάτι που διαταράσει τις καλές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ερευνητικέ δραστηριότητες δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι έγιναν παράνομες τέτοιες πράξεις στην βορειοανατολική Πολωνία και έγιναν εκεί παραδόσεις. Είναι προφανές ότι τέτοιες δραστηριότητες της CIA θα μπορούσαν να είχαν λάβει χώρα μόνο υπό την αιγίδα και την ευλογία ε, των διαφόρων αυτών χωρών που αναφέρονται. Αυτό σημαίνει ότι ανώτατοι αξιωματούχοι συμμετείχαν στις πράξεις αυτές, στις παράνομες δραστηριότητε της CIA. Και αν δεν απολογηθούν και αν δεν πούν ότι αυτό είναι πραγματικό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι δυνάμεις ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρελθόν συμμετείχαν στις δραστηριότητε του Πινοσέ. Δεν πρέπει να επαναληφθεί. Είναι συνάδελφος Μπρόνς. Η παράνομη κράτηση δεν είναι κάτι εσφαλμένο από μόνο του, είναι παράνομο. Δεν υπάρχουν αρχεία πραγματικά, οπότε διευκολύνεται η κακομεταχείριση του κρατουμένου. Δεν χρειάζεται να πω ότι τα βασανιστήρια ποτέ δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ηθικά. Όμω, αν δεν πείθονται με ηθικά επιχειρήματα κάποιοι, να υπενθυμίσουμε ότι είναι αναποτελεσματικά τα βασανιστήρια. Διότι οι πληροφορίε που αποκτώνται δεν είναι αξιόπιστε. Και η αξία προπαγάνδας για του τρομοκράτε που έχουν υποφέρει είναι τεράστια. Οι πολιτικοί ηγέτε σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τι πράξει του. Και κάποιοι φαίνεται ότι πράγματι θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Όμω αυτοί, όπω και οι κρατούμενοι τρομοκράτε, πρέπει να θεωρούνται ε, καταρχήν ε, αθώοι σε οποιαδήποτε δίκη. Πλήρε δικαστικέ έρευνε είμαι πεισμένο θα πρέπει να γίνουν στι διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Όμω είμαι αντίθετο τη νομοθεσία που ζητά το ψήφισμα. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει γενικά την εξουσία, ούτω ώστε να, θέσει τις, να ελέγξει τι υπηρεσίε ασφαλεία των 100 μελών. Αυτό είναι θέμα που αφορά το δικαστικό σώμα και τι διάφορε αρμόδιε αρχέ των κατών μελών. Ευχαριστώ. πολύ κύριε καλώ στο βήμα την ε, Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ εξ ονόματος της Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, εξ αρχής η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά σε αυτό το ζήτημα ήταν η εξής. Πρώτον, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται ε, σεβόμενη πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει να βρεθεί η αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή, και τρίτον, ότι θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να υπάρξει ε, πρόληψη και να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους πράγματα στο μέλλον. Η κυρία εισηγήτρια γνωρίζει, το γνωρίζει αυτό, διότι της έχουμε απαντήσει σε πολλές επιστολές μας. Η πρώτη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συντάχθηκε το 2006 από τους συνοδέλφους μου Φρατίνη Μπαρό, ο Μάλστρομ και στη συνέχεια και από εμένα. Και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στα κράτη-μέλη, ώστε όλη η αλήθεια να έρθει στο φως. Επίσης, θα συναντηθώ με τον κύριο Σταύρο Λαμπρινίδη, τον ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα συνεργαστούμε για να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ως προς τις ενδιαφερόμενες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω ότι έχουμε έναν μόνιμο διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία. Και ε, σύμφωνα με όλη το, σύνολο του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τη σύμβαση για κατά των βασανιστερίων. Πολύ συχνά ε, στο διάλογο που έχουμε με όλες τις τρίτες χώρες ε, θέτουμε τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα βασανιστήρια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να σας πω ότι η κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των ανθρώπων από την ε, κατεξαναγκασμό ε, εξαφάνιση υπάρχει και εμείς έχουμε δηλώσει την επιθυμία μας να έχουμε κυρώσει αυτή τη σύμβαση σε στο πλαίσιο του ICCPR μέχρι το 2015. Τέθηκε ένα ερώτημα εδώ στην Ολομέλεια. Θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Θέλω να απαντήσω ξεκάθαρα όχι. Δεν θα, Δεν θα ξανασυμβεί γιατί τώρα μιλούμε με δυνατή φωνή. Δεν θα ξανασυμβεί διότι το Κοινοβούλιο δεν ε, σταματά να ασκεί πίεση. Και δεν θα ξανασυμβεί, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας της κοινωνίας μας από τη μία και των δικαιωμάτων των πολιτών μας από την άλλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος όπου επικρατεί το κράτος δικαίου, θα πρέπει να κάνουμε το παν, να χυθεί άπλετο φως στα γεγονότα του παρελθόντος, ώστε τέτοιου είδους συμβάντα να μην επαναληφθούν πολύ κυρία Επίτροπε. Ε, η ζήτηση ολοκληρώνεται με την εισηγήτρια κυρία Φλότ. Έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ όλους εκείνους που παρενέβησαν στη συζήτηση θέλοντας να υποστηρίξουν τη δουλειά που έγινε μακρόπνοη εργασία σε ένα χρόνο έχουμε ραντεβού όπως είπα στην αγωγή εδώ μετά από ένα χρόνο μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στα κράτη-μέλη. Βεβαίως δεν είμαστε δικαστικοί εδώ. Ε, δεν έχουμε πλήρες αποδείξεις. Ξέρω μόνο από τη Ρουμανία ότι έγινε στη Γερουσία μια έρευνα, το ανέφερα, αλλά ξέρω ότι διάφορες εικασίες, νέες πτήσεις που συνδέουν Ρουμανία με Λιθουανία, ε, αναφέρθηκαν το Eurocontrol και σε μια καταγγελία κατά της Ρουμανίας στο Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργήθηκε φάκελος από τον Επίτροπο Ανερμπέργκ, τον Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν ξέρουμε ακόμα τα πορίσμα τη έρευνας. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε συγκεκριμένη χώρα. Επέμεναν πολλοί διάφοροι συναδέλφοι επέμειναν επί συλλογικής ευθύνης που έχουμε. Τι συμβαίνει. Κάθε χώρα έχει ένα κομμάτι της αλήθειας. Και χρειαζόμαστε, ζητούμε κάθε χώρα να κάνει τις καλύτερες δυνατές έρευνες για να ρίξουμε φως στο σύστημα. Διότι πρόκειται για ένα σύστημα. Δεν αναφέρουμε συγκεκριμένη χώρα, δεν κατοικούμε συγκεκριμένη χώρα, είναι σαφές. Κανείς δεν το αρνείται ότι στη Ρουμανία μια νέα έρευνα δικαστική θα πρέπει να ξεκινήσει. Διότι τα στοιχεία που δεν είναι αποδείξεις, δεν είμαστε δικαστές, τα στοιχεία είναι αρκετά σημαντικά, ούτω ώστε να δικαιολογηθεί άνοιγμα εκ νέου μια έρευνα. Η έκθεση ζητά κάτι διαφορετικό. Ζητά η έκθεση από τις χώρες να ξεκινήσουν έρευνες. και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αναφέρει ότι ένα κομμάτι της αλήθειας έχει κάθε χώρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα μέσα, την εξουσία και το καθήκον, την υποχρέωση να φροντίσει τους, ώστε αυτό το κομμάτι της αλήθειας να είναι σαφές να δοθεί σε άλλες χώρες, να διαφωτιστούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να κάνετε πάρα πολλά. Υπενθυμίστηκαν οι κανόνες. Είσαστε στεναροί, σταθεροί, αυστηροί. Μιλάτε πολύ συχνά για την παραβίαση των θεμελιών δικαιωμάτων στα πλαίσια της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου αλλά στην πλαίσια αυτών των προφανών τεραστίων παραβιάσεων που δεν έχουν διαφωτιστεί θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία για τις παραβιάσεις. Όσον αφορά το θέμα που μας αφορά, μπορείτε να συναθρήσετε τους ε, διαφόρους εισαγγελείς. Μπορείτε να μεταφράσετε όλα τα χρήσιμα έγγραφα. Μπορείτε να μαζέψετε τις πληροφορίες, να τις δώσετε στα κράτη για να βοηθήσετε τις χώρες να διεξαγάγουν τις έρευνες και στην επιστολή που χαίρομαι θα στείλετε σε κάθε χώρα θα πρέπει όλα τα λένε στοιχεία να αναφέρονται ε, κυρίως μέσω της αναλύσεως που έγινε από τα στοιχεία του Eurocontrol για τις πτήσεις. Θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά σε ένα χρόνο και ελπίζω μόνη μου την καρδιά ότι σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να δώσουμε ραντεβού και να τρέξουμε συμπεράσματα. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ την ε, εισηγήτρια, την κυρία Φλότ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση κηρύσσεται περιομένη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τώρα το επόμενο σημείο στη μίλησια διάταξη είναι παρεμβάσει ε, διάρκεια ενός λεπτού. Ε, απευθύνω θερμή παράκληση να τηρούμε τον χρόνο του ενός λεπτού. Ε, επιτρέψτε μου να πω ότι θα είμαι αυστηρός ε, σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις θα είναι πράγματι ε, ενός λεπτού γιατί μας πιέζει το χρονοδιάγραμμα εργασιών. Δίνω το λόγο στην ε, συνάδελφο κυρία Μαρία Πατράου Νέβες. Κύριε Πρόεδρε, το Σεπτέμβριο πολλοί κάνουν